μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Με την έννοια του άρθρου 198 του κανονισμού, η διάσκεψη των Προέδρων έλαβε ένα αίτημα από 283 μέλη του Κοινοβουλίου να συσταθεί μια διερευνητική επιτροπή για, τις, για τη μέτρηση των εκπομπών των αυτοκινήτων. Και η διάσκεψη των Προέδρων έλαβε υπόψη της ότι το έτοιμο αυτό υποβλήθηκε όπως προβλέπεται. Ε, αποφάσισε ε, πάνω από ένα τέταρτο μελών να ληφθεί απόφαση στην Ολομέλεια όσον αφορά τη σύσταση διερευνητικής ε, επιτροπής, το πώς θα απαρτίζεται η επιτροπή αυτή και η διάρκεια της εντολής της. Η πρόταση σχετικά με την απόφαση που φέρει και την ε, ε, απόφαση Β8 ε, Παύλα 1424 του 2015 αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και θα ψηφίσουμε αύριο γι' αυτό οι τροπολογίες στην πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με την αριθμητική σύσταση, το πώς θα μετέχουν δηλαδή ε, στην Επιτροπή αυτή, η πρόταση μπορεί να καταδεθεί μέχρι τις 8 σήμερα το βράδυ. Θα ψηφίσουμε ε, σχετικά με την σύσταση αυτής της Επιτροπής, το ποιος θα επναπαρτίζει στις 19 Ιανουαρίου. Σήμερα λοιπόν ε, η ημερήσια διάταξη, μισό λεπτό, έχετε το λόγο, ο κύριος Μαριάς διαδικαστικό. Άκουσα την ανακοίνωσή σας ότι έχουμε δικαίωμα ό,τι είναι να το προτείνουμε μέχρι τις 8 η ώρα. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι μια διαδικασία δημοκρατική, διότι όπως βλέπετε εδώ είναι ελάχιστοι συνάδελφοι, ο χρόνος που δίνεται είναι μία ώρα και αντιλαμβάνομαι ότι αυτές δεν είναι διαδικασίες για ένα κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει άνεση χρόνου, αλλά το να μας λέτε ότι μέσα σε μία ώρα θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση. την ώρα που δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή θεωρώ ότι πρέπει να το ξαναδείτε αυτό. Κοιτάξτε, εμεί ε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συζήτηση από αυτού, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, λόγω του κανονισμού, των όσων προβλέπει ο κανονισμό. Αυτή η απόφαση ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων και η διάσκεψη των Προέδρων καθόρισε και το τι θα ισχύει για την κατάθεση των τροπολογιών. Όσον αφορά την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λάβουμε υπόψη μας αυτή την απόφαση. Δεν μπορούμε τώρα δυστυχώς να κάνουμε συζήτηση. Τώρα, ε, προβλέπετε ότι ε, θα ακολουθήσει συζήτηση για θέματα ασφαλείας. Ε, πρόκειται και για την 21η επέτειο από την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης, η Συμφωνία του Ντέιτον. Το λόγο έχει ο κύριος